εταιρική ευθύνη και στην υφόρο ανάπτυξη της Διεθνής εμπορικής συμφωνίας Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεζίρ. Κλείνει η συζήτηση του θέματος αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 η ώρα, αν θέλει ο Θεός. Ακολουθούμε στο τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης, που είναι η προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για τις περιπτώσεις αντι-dumping την τωρινή κατάσταση και τις προοπτικές είναι μια προφορική ερώτηση από το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές, φιλελεύθερους, γκούε, πράσινους και συντηρητικούς. Β70562 κάθετος 10 συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντάκτες αυτής της προφορικής ερώτησης. Δύο λεπτά κύριος Κασπάρη. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, το anti-dumping παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον κόσμο μας και νομίζω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται για πρώτη ξιονισμό, προστατευτισμό, αλλά μια σωστή εφαρμογή τη αρχή του αντι-dumping. Ξέρουμε ότι είναι στρεβλωτικέ οι κρατικέ επιδοτήσει σε πολλέ περιπτώσει. Θα πρέπει εμεί να έχουμε τον τρόπο να προστατευτούμε όταν υπάρχουν προϊόντα dumping τα οποία έρχονται στην αγορά, τα οποία πολλούνται κάτω του κόστου. Κύριε Κασπάρη, ποια διερμηνία δεν λειτουργεί. Εντάξει, όλα, όλα είναι εντάξει. Συγγνώμη. Πρόκειται για προϊόντα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, για τα οποία οι επιχειρήσει θα φέρουν φτηνότερα στην αγορά από ότι στο κόστο, στην τιμή του κόστου, ένα τρόπο να σπρώξουν στην άβυσο του άλλου ανταγωνιστέ του κάτι το οποίο είναι αφέμητο. Θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν αν έχει εμπειρίες αυτού του είδους και αν υπάρχει κάποια γνώση και από την πλευρά της Κομισιόν και του Συμβουλίου αν υπάρχουν ξένες κυβερνήσεις οι οποίες ακολουθούν τέτοιες εμπορικές ε, πρακτικές. Αν ξένες κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ξένες κυβερνήσεις κάνουν εμπορικές ενέργειες οι οποίες βρίσκονται στα πλαίσια του dumping και μας έχουν οδηγήσει σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Νομίζω ότι αυτό θέλω να το γνωρίσω γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες γεμάτες από ανησυχίες έχουν έρθει σε μένα και με έχουν ερωτήσει τι γίνεται και επίσης μου ζητήσαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μάθω ποια είναι η άποψη της περίπτωσης ε, από την πλευρά της Κομισιόν. Πολλές φορές η επιβολή δασμών εμποδίζει τις δικές μας επιχειρήσεις σε χώρες της Ασίας και αλλού να πολλούν τα προϊόντα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων όπως τη βλέπει η Κομισιά. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Πάλι για δύο λεπτά. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μουρέα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Πίτρουπε, θα ήθελα τώρα να διευκρινίσω στο βαθμό του δυνατού ποια είναι η θέση της Επιτροπής ε, <clears throat> Εξωτερικών Υποθέσεων για τα θεματα αντι anti-dumping και προστασίας από τέτοιες αθέμητες ε, πρακτικές. Είναι γεγονός ότι η Κομισιόν σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή της έλεγε ότι δεσμεύεται να φιλελευθερωποιήσει το εμπόριο στα πλαίσια του θεμητού ανταγωνισμού μεταξύ εγχωρίων και ξένων παραγωγών. Πρέπει όμως να προστατεύονται οι παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από στρεβλόψη του διεθνούς εμπορίου και να εφαρμόζονται αμυντικά όπλα <clears throat> αντιντάμπινγκ μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αλλά πέραν αυτής της θετικής νομικής πρόσας, το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι πράγματι ε, εφικτή αυτή η στόχη οι οποίοι επιδιώκονται. Είναι δυνατόν λοιπόν η πρόσφατη πρόταση του Συμβουλίου για τον έλεγχο στα κάτι μέλη των πράξεων της Κομισιόν μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα μέτρα προστασίας σε εμπορικό επίπεδο anti-dumping αυτές στρέφονται κατά της ανάγκης εγγύησης του ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα anti-dumping. Προβλέπει Συγκεκριμένα η πρόταση του Συμβουλίου εξαιρέσεις γενικές στα θέματα της επιτροπολογίας που εμποδίζουν, κολλησιεργούν, πολιτικοποιούν και εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά που τελικά είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν. Και επίσης θα ήθελα να πω το εξής, στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται ότι θα υπάρξει ο εξυγχρονισμός και η επικαιροποίηση των εργαλείων μας για εμπορική άμυνα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Κατά πόσο εφόσον η Κομισιόν δεν αντιτίθεται στη θέση του Συμβουλίου για την διαδικασία που αφορά τα εμπορικά αντίμετρα, τι εγγυήσεις μπορεί να μας δώσει η Κομισιόν ότι όταν, έχει, όταν έρθει η στιγμή της αναθεώρησης αυτών των μέτρων θα μπορέσει να υψώσει το ανάστημά της έναντι των ίδιων αυτών κρατών μερών που θέλουν να εμποδίσουν τη λήψη αντιμέτρων κατά του ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Μουρέιρα, ακολουθεί για δύο μισή λεπτά ο κύριος Ρινάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε λίγοι απόψε που για να μιλήσουμε για το αντι που όμως είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάνε πολλοί στις χώρες μας. Νομίζω ότι στα θέματα του διεθνούς εμπορίου δεν υπάρχει θέμα πιο πολύ στο επίκεντρο των ε, ενδιαφέροντων των επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνδικάτων, των καταναλωτών από το dumping. Εμείς ζητάμε το θέμα αυτό, γιατί είναι η αντιπαράθεση με το ντάμπινγκ είναι καθημερινό ψωμί στον παραγωγικό μας τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται, κάνει την προσπάθειά τη, ε, κάνει το καθήκον τη όσον αφορά τι πρωτοβουλίες αντι-dumping, αλλά εμείς ε, ζητάμε μια δράση η οποία να εμπνέεται από τις κάτω θεαρχές. Πρώτα απ' όλα αδιαφάνεια όσον αφορά τη δράση πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών, των κριτηρίων αξιολογήσεως που υιοθετούνται και των αποτελεσμάτων. Και μετά η επικοινωνία, η στατηγική επικοινωνία, ούτω ώστε οι δράσει αντι-dumping τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να είναι ένα στοιχείο διαβεβαίωσης, ε, καθεσυχασμού αν θέλετε για τους επιχειρηματίες μας και για τους εργαζομένους μας. Δεύτερον, υπάρχει ένα περιθώριο διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διαδικασία του dumping. Αυτό ανήκει στην κοινή λογική. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι ξεπερνά αυτή τη δυνατότητα διάκριση όσον αφορά τι αποφάσει που λαμβάνονται. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην φάση αυτή μετά τη Λισαβόνα και θα πρέπει να ενημερώνεται και να συμμετέχει περισσότερο σε αυτές τις διαδικασίες. νομίζω ότι υπάρχει ένα είδο κοπόσεω από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το να μπορεί να αναγνωρίσει πλήρω το ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Αν και αναφυσβήτα γίνονται πάρα πολλέ προσπάθειε και ευχαριστούμε για αυτό τον κύριο Επίτροπο, αλλά σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει περισσότερο βάρο όσον αφορά το κεφάλαιο αυτό του αντι-dumping ε, το θέμα του διαλόγου με την κοινωνία ε, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει μόνο ε, και ανακούει του ε, φορεί και του εκπροσώπου των διαφόρων φορέων και για το αντι και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταγράψει τις νέες απαιτήσει που υπάρχουν όσον αφορά τις αποκριστικές αρμοδιότητες για το διεθνές εμπόριο που ε, απορρέουν από τη Λισαβόνα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλο, είναι σαφέ ότι για μα το anti θα πρέπει να αποτελεί ένα τμήμα στρατηγική εμπορική που θα είναι συνεκτική, μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα εμπνέεται από τα κριτήρια της, του θεμητού ε, ανταγωνισμού και του ανοίγματο. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε το κεφάλι ψηλά από εδώ και πέρα. Σα ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Ρενάλντι. Επόμενο για δύο λεπτά είναι ο συνάδελφο Σλούτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορούμε να δούμε τώρα τι επιπτώσεις. Κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άδραξε την ευκαιρία για να τροποποιήσει το 2007 αυτό το μέσο ε, προστασία ε, στα πλαίσια του Global Europe. Αυτό ήταν ο στόχο. εξάλλου. Επίσης, Υπάρχει το θέμα της Λισαβόνας και ποιες διαδικασίες πρέπει να έχουμε. Κάποιες που έχουν ίσως δεν είναι πλέον ενδεδειγμένες οι πράσινοι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο κάτω-κάτω της γραφής. Ε, ε δεν θα είναι, υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής άμα είναι δίκαιοι και διαφανείς και σαφείς οι κανόνες. Θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε τα συμφέροντα των παραγωγών. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα συμφέροντα των καταναλωτών όπως είπε και ο κύριος Κασπάρη, θέλουμε να σταματήσουμε το dumping ε, αλλά υπολογίζοντας το πραγματικό κόστος παραγωγής. Το πραγματικό κόστος πρέπει να καλύπτει όμως και το περιβαλλοντικό dumping. Ε, και ε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών επιδοτήσει. Ε, δηλαδή είτε μιλάμε για την οικονομία είτε για το περιβάλλον. Πρέπει να υπολογίσουμε το κόστο και να το συνυπολογίσουμε και αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε περίπτωση dumping. Τώρα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την εμπορική πολιτική για να επιτύχουμε άλλου στόχου. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέτρα αντι-dumping στα πλαίσια του συστήματο εμπορία ρήπων για να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ε, υπάρχουν εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες εταιρείες με τέσσερα διαφορετικά κριτήρια σχετικά με το πώς μπορούν να εξαιρεθούν από το σύστημα εμπορίας ρήπων ή να έχουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Για ποια διαδικασία μιλάμε όταν ε, ε, πλήττονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, από αθέμητο ανταγωνισμό, επειδή άλλες χώρες δεν έχουν τα ίδια πρότυπα και στους κανόνες. Σας ευχαριστούμε κύριε Σλάιτερ. Δύο λεπτά ο κύριος Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ήδη από την προηγούμενη συζήτηση έχουμε τονίσει την ανάγκη η εμπορική πολιτική να εμβαπτιστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να μπορέσει να συνάδει με το διεθνέ δίκαιο, με την προστασία του περιβάλλοντο, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη θα πρέπει επομένω να λειτουργήσουν με τον αντίστοιχο τρόπο στον ΠΟΕ. Εμεί έχουμε επικρίνει σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρική μα ομάδα τον τρόπο με τον οποίο δρά στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προασπίσει και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ε, εργαζόμενους έναντι των εξωτερικών μορφών αθέμητου ανταγωνισμού. Θα πρέπει να είμαστε σαφέστεροι λοιπόν σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής και να αγωνιστούμε και κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ και του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ που όπως είπαν οι συνάδελφοι μειώνει το κόστος, <clears throat> το φαινομενικό κόστος παραγωγής. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο στην Ευρώπη λόγω αυτού του αθέμητου ανταγωνισμού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να έχουμε ένα ορισμό του πραγματικού κόστους μέσα από ένα, ε, ένα ορισμό ο οποίος είναι αντικειμενικού χαρακτήρα και δεν βασίζεται σε αυθαίρετες επιλογές. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάθε συμφέρον να προστατευτούν από το αντιτάμπινγκ και όμως δεν τη χάνουν της ίδιας προστασίας όποιο πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους ε, εργαζόμενους στην Ευρώπη να έχουν την απαραίτητη υποστήριξη από την Κομισιόν. Θα ήθελε η Κομισιόν λοιπόν να υλοποιήσει μια τέτοια προσέγγιση και να δράσει σε περιπτώσεις όπως της Σανγκομπέν ε, στο παρελθόν. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τέτοιες εμπορικές πρακτικές θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την απαραίτητη ευρωστία και εκπροσώπηση για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Ο κύριος Στούρδη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε από την αρχή της οικονομικής ύφεση. επανειλημμένα υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ακολουθήσει προστατευτικές πολιτικές αλλά να προωθήσει την απελευθέρωση του εμπορίου και εσείς ήσασταν υπέρ αυτής να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες να δημιουργήσει θέλητρα για επενδύσεις στην Ευρώπη. Συμφωνώ ότι τα μέτρα αντι-dumping πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητα. Το πρόβλημα όμως βέβαια είναι ότι αν τα χρησιμοποιούν χρησιμοποιείται ως προστατευτικά μέτρα. Ε, μόνο και μόνο ο αριθμός των ερευνών αντι-dumping που γίνονται αυτή τη στιγμή υποδεικνύει ότι ε, χρησιμοποιείται για διαφορετικό στόχο αυτό το μέτρο αντι-dumping. Ζητώ συγγνώμη, πριν από τέσσερι εβδομάδε σα μιλούσα ε, για ένα πρόβλημα με μια εταιρεία ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Βέλγιο και τελικά το έλυσαν μόνοι του το πρόβλημα. και ε, αλλά δεν κινήσατε την ε, νομοθεσία περί αντι-dumping κατά αυτές τις εταιρείες. Ήταν μια βελγική και μια κινέζικη εταιρεία. Τέλος πάντων συνεργάστηκαν ούτω ώστε να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργήσουν ευκαιρίε. Ε, θα σα δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη έχουμε ένα θέμα με το με το γυαλί ε, και έχουμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ε, με τις ίνες γυαλιού είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το προϊόν, ε, χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές για διάφορα προϊόντα και υπήρξε μια αντίστοιχη περίπτωση όπου δεν χρειάστηκε να παρέμβετε. Ο προ-προ κάτοχό σας επίσης εφάρμοσε για τα λοιπάσματα τέτοια πολιτική αντι-dumping και κλειδονίστηκε ο κλάδος ε, και ως προς τους προμηθευτές και ως προς την παραγωγή ε, και ως προς το κόστος των προϊόντων έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις αντι-dumping κατά 173%. Μα για ποιο λόγο αφήστε τις αγορές σε ήσυχες. Εσείς ειδικά θα έπρεπε να ξεφορτωθείτε αυτό τον προστατευτισμό ε, που σοβεί στην Ευρώπη. Περιμένω με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας, Επίτροπε Ντεγκού. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Στέρντι ο Επίτροπος Δεγκούχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψή μας ότι η προάσπιση των Ευρωπαίων παραγωγών έναντι εξωτερικών στρεβλώσεων του εμπορίου θα πρέπει να θεωρείται ένα παράγραπτο ε, συστατικό στοιχείο μιας ε, εισοδικία στρατηγική εμπόριου. Νομίζω ότι οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά και αντικειμενικά στοιχεία και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι έχουμε ένα από τα πιο εισοδίκια και αποτελεσματικά συστήματα άμυνα στον κόσμο κατά του ντάμπινγκ. Υπάρχουν φυσικά πολλά συμφέροντα που εμπλέκονται στο ντάμπινγκ και στην παροχή κρατικών επιδοτήσεων και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Αλλά μπορώ να σας πω ότι η διαδικασία αυτή είναι διάφανη και αποτελεσματική και βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Αναγνωρίζω ότι πρόσφατα τρίτες πλευρές έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν τη λήψη απόφασης ε, πιέζοντας τα, τις επιχειρήσεις οι οποίες διαμαρτύρονται ή ακόμα και κράτη-μέλη τα οποία, στα οποία εργάζονται αυτές οι εταιρείες. Εμείς καταδικάζουμε στεναρά αυτές τις πράξεις. στα πλαίσια αυτά η εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας δίδει μια δυνατότητα να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο αριθμός των περιπτώσεων αντι-dumping εξακολουθεί να μένει σταθερό σε συνάρτηση του χρόνου. Κύριε Στέρντι, δεν ανεβαίνουν λοιπόν οι αριθμοί αυτών των περιπτώσεων. Έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε οποιαδήποτε αισθητή αύξηση που μπορούσε να είχε προκληθεί από την παγκόσμια ύφεση και εξασφαλίσουμε ότι το dumping δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ή μάλλον η διαδικασία αντι-dumping δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστατευτικούς λόγους. Οι στατιστικές δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιπτώσεις αυτές είναι μικρότερες από τις τους κύριους εμπορικούς φορείς του κόσμου. Η Κίνα παραμένει ο σημαντικότερος χώρος όπου υπάρχουν προβλήματα dumping και είναι το 1 τρίτο των περιπτώσεων που έχει αναλάβει δράση ε, ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Κίνας. Ο κύριος Στέρτ διέθεσε και ένα ερώτημα στην, ε, περίπτωση, λεγόμενη περίπτωση Modem διαμορφωτών διαμορφωτων όπου κοίταξε η Κομισιόν θέματα dumping, επιδοτήσεως και επί τη βάση <clears throat> καταγγελιών μιας ε, ανταγωνίστριας εταιρείας. Βάσει του βασικού κανονισμού, οι παραπονούμενοι μπορούν να αποσύρουν τα παραπονά τους. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, όταν αποσυρθεί η καταγγελία, μπορεί να τερματιστεί εκτός αν ο τερματισμός της διαδικασίας δεν θα είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς εξετάζουμε τώρα τις συνέπειες της απόσυρσης της καταγγελίας. Στο παρελθόν η Κομισιόν έχει δεχτεί τέτοιες ε, αποσύρσεις καταγγελιών και έχει τερματίσει την έρευνα χωρίς περαιτέρω μέτρα. Στην τρίτη περίπτωση, οι διασφαλίσεις για μια καταγγελία η οποία έγινε από μια κυβέρνηση που τυχαίνει να είναι και η βελική κυβέρνηση, είναι κάπως διαφορετική διαδικασία. Η αντίστοιχη εταιρεία έχει πληροφορήσει την ε, Κομισιόν ότι ζήτησε η βελική κυβέρνηση να αποσύρει την αίτηση για μέτρα διασφάλισης. Αλλά η βελική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα πληροφορήσει την Κομισιόν εάν θα συμμορφωθεί με την αίτηση αυτή που έχει υποβάλει η εταιρεία αυτή. Επομένως περιμένουμε να δούμε, να δούμε ποια είναι η θέση της φελικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεχίζουν λοιπόν σε ευρύτερο επίπεδο τα εργαλεία προστασίας του εμπορίου υπάρχουν για εύλογους λόγους. Αν δεν υπάρχουν διεθνείς κανόνες για το εμπόριο και δεν υπάρχουν πλήρεις αγορές, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε την παραγωγή μας έναντι στρεβλωτικών μορφών αθέμητου ανταγωνισμού. Προσπαθούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την χρήση ε, χρονικών ορίων, έχουμε και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για του εξαγωγεί. Και όλα αυτά έχουν σαν στόχο να είναι ισοδίκια και να είναι προ το όφελο όλων των εμπλεκομένων κοινωνικών, εμπορικών μάλλον φορέων. Οι διεθνεί κανόνε για την εμπορική άμυνα είναι υπό αναδιαπραγμάτευση στον ΠΟΕ. Η θέση Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική. Θέλουμε να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων, ενώ συγχρόνω προστατεύουμε τι επιχειρήσει μα από προστατευτικέ ενέργειε άλλων. Οι διαπραγματεύσει λοιπόν στα πλαίσια του ΠΟΕ και οι αλλαγέ οι οποίε έχουν προκύψει από τι συνθήκε τη Λισαβόνα είναι σημαντικέ για την αναθεώρηση, για οποιαδήποτε αναθεώρηση των κανόνων μα που θα μπορούσαμε να πράξουμε. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τα εργαλεία για την προστασία του εμπορίου είναι πάρα πολύ σημαντικά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ό,τι αφορά το κόστο και την πολυπλοκότητά του. Υπάρχει μια προσπάθεια να μειώσουμε στι έρευνε αντι-dumping το διοικητικό άχθο. Γι' αυτό η Κομισιόν ξεκινήσει να ερευνά τι ειδικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίε επιχειρήσει όταν έχουν να αντιμετωπισουν περιπτώσει περιπτώσεις αντι-dumping και τι δυνατότητε να ανακουφίσουμε αυτό το άχθο. Σε ό,τι αφορά τώρα τι θεσμικέ πλευρέ, θα έχετε σημειώσει ίσω ότι οι πρώτε επιτροπολογίε που υπερβλήθη από την Κομισιόν το Μάρτιο <clears throat> προβλέπει να υπάρχει πλήρης πληροφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις διαδικασίες αυτές επιτροπολογίε. Η Κομισιόν επίσης θα δώσει πληροφορίες για τα μέτρα βάσει των οποίων προβλέπεται η γνωμοδότηση πριν από την τελική έγκριση του μέτρου αυτού από την Κομισιόν. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πάρει περαιτέρω πληροφορίες από την Κομισιόν εφόσον το επιθυμήσει. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω και πάλι ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να κάνει μια πρόταση για την ευθυγράμμιση των εργαλείων προστασία του εμπορίου με το νέο σύστημα ελέγχου των κατεχώρησης ε, πράξεων. Είναι το λεγόμενο λεωφορείο του εμπορίου. Αλλά η συζήτηση των θεσμικών οργάνων για το σύνολο των εφαρμοστικών πράξεων συνεχίζεται. Η Κομισιόν προσεκτικά παρακολουθεί τη συζήτηση και εκτιμά επί τη βάση των επαφών με τα άλλα θεσμικά όργανα πότε θα πρέπει να αναλαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Αλλά αυτό γίνεται όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Ανεφέρθη και από τον πρόεδρο Μορέιρα το θέμα της επιτροπολογίας και δεν να είμαι πάρα πολύ σαφής. <clears throat> Δεν βλέπω αποχρόντα λόγο και κανένα στοιχείο στη συνθήκη της Λισαβόνας που θα οδηγούσε σε μια ειδική αντιμετώπιση της επιτροπολογίας όταν πρόκειται για εμπορικά θέματα. Δεν θα συμφωνήσουμε λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια ειδική μεταχείριση. Φυσικά η απόφαση αυτή εξαρτάται και από το Συμβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και η Κομισιόν θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο και ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική πλειοψηφία που θα τροποποιούσε, που θα απέτυχε τη θέση Κομισιόν. Αυτό όμως δεν είναι αποδεκτό για μένα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα αμυντικά του εμπορίου εργαλεία έναντι τρίτων χωρών, έχουμε δει πράγματι από την αρχή της οικονομικής κρίσης μια μεγαλύτερη χρήση αυτών των εργαλείων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά τις αμυντικές δράσεις τρίτων χωρών και παίρνουμε δράση όταν αυτό είναι απαραίτητο. Έχουμε λοιπόν παρακολούθηση ε, διαδικασίες κατά Ευρωπαίων εξαγωγέων και καταγγελίες των ΠΟΕ. Σε πολλές περιπτώσεις η δράση της Κομισιόν οδηγεί στην περάτωση της ε, έρευνας χωρίς την εφαρμογή μέτρων. Άλλες φορές αυτές οι παρεμβάσεις οδηγούν σε χαμηλότερες κυρώσεις για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Και υπήρχε επίσης υπήρχε το θέμα αυτό για τα αντίμετρα κατά τρίτων χωρών που ασκούν αθέμητες πιέσεις στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Έχουμε λάβει αναφορές σε σχέση με τα θέματα αυτά από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά τις κρατάμε ανώνυμες για να προστατεύσουμε τους αθώους στην περίπτωση Φάστρες που αφορούσε την Κίνα. Η Κίνα το έθεσε το θέμα αυτό στο πάνελ του ΠΟΕ για την ε, ρύθμιση διαφορών. Μας υποστήριξε το πάνελ, αλλά δεν έχουμε πει ποιες ήταν οι εταιρείε γιατί πρέπει να τις προστατεύσουμε. Και δύο τελευταία ερωτήματα για το αν θα υπάρξει αναθεώρηση των εργαλείων για την προστασία κατά του τάμπινγκ. Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό γιατί πιστεύω εκ βάθου καρδίας ότι δεν είναι απαραίτητο καταρχήν. Είναι πολύ μεγάλο το έργο που πρέπει να κάνουμε στα επίπεδα εμπορίου του επόμενου χρόνου. Και δεν θέλω να ξεκινήσω και πάλι κάποιες συζητήσεις μέσα σε μια τέτοια διαδικασία αναθεώρησης. Θα το εξετάσουμε αυτό μόνο όταν τελειώσει ο γύρος της Ντόχα. Υπάρχει επίσης ένα ερώτημα πιο συγκεκριμένο που ετέθη από ένα πράσινο μέλος. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά σας. Α, ο κύριος Σλίτερ. Είσαστε ένας πολύ, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του Μεσαίωνα, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα του κυρίου Σλούτερ. Όπως ξέρουμε αυτές τις περιπτώσεις αντι-dumping υποβάλλονται από εταιρείε επί τη βάση καταγγελιών εταιριών. Αν μια εταιρεία έθετε το θέμα το οποίο εσείς αναφέρατε προηγουμένως για την διαρροή άνθρακος, δηλαδή με την κατάσταση επιχειρήσεων, τότε η Κομισιόν αυθορή και παραχρήμα θα προέβαινε σε έρευνες και θα έβλεπε αν αυτό πρέπει να οδηγήσει σε αντισταθμιστικά μέτρα. Δεν αποκλείεται από την εμβέλεια των επιχειρημάτων που μπορούμε να εξετάσουμε. Εμείς θα εξετάζαμε λοιπόν τα επιχειρήματα της εταιρείας. Αν μια εταιρεία λοιπόν έθετε το θέμα αυτό θα το εξετάζαμε. Ε, ευχαριστούμε τα μάλα κύριε Επίτροπε. Κύριε Στέρντι, δεν μπορούμε να διακόπτουμε τους επιτρόπους με μπλε κάρτες, ούτε κάνουμε πορτοκαλί. Ακολουθούν οι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Μοσχαρδίνη, για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, το αντιντάμπινγκ που αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για άμυνα για την σωστή εφαρμογή του εμπορίου στην Ευρώπη μπορεί χρειάζεται σαφεί κανόνε και εφαρμόσιμου κανόνε εντό τη νέα επιτροπολογία. Η συνθήκη τη Λισαβόνα λέει σαφώ ότι οι εκτελεστικέ πράξει είναι στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο. Έχει την εξουσία να ελέγχει την λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συμβιβασμό που εξετάζεται σήμερα αφαιρεί εκ των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο το ρόλο που η Λισαβόνα του είχε αναθέσει και θα μπορούσε έτσι να δημιουργηθεί ένα νέο δημοκρατικό έλλειμμα εντός ε, των θεσμών θεσμικών οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, δεν καταλαβαίνουμε και απορρίπτουμε την πρόταση να υπάρχει διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των μέτρων Αντιμετώπιση που εισάγει στοιχεία διακριτικής μεταχείρισης, πολιτικής χρειάς και νομικής αβεβαιότητας σε διαδικασίες που μέχρι τώρα έπρεπε να προστατεύονται θεμητά συμφέροντα επιχειρήσεων που ευλάπτονται από αθέμητο ανταγωνισμό. Σε σοβαρή περίοδο περνάμε οικονομικής κρίσεως όπως αυτή, ε, θεωρούμε ότι θα ήταν παράλογο ε, και αυτοτραυματικό ε, να καθιστούμε περίπλοκο και περίπλοκη και μη αποτελεσματική τη διαδικασία την dumping. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα της προτάσεως που υπευλήθη εάν δεν τροποποιηθεί. Και καλούμε να αναλάβει τις ευθύν, να αναλάβουν τις ευθύνες τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη τον οποίο το κοινό συμφέρον θα έπρεπε να είναι η εγγύηση μεγαλύτερης ανάπτυξης και ανάπτυξη μπορεί να γίνει μόνο παρουσία κανόνων που αποφεύγουν τη στρέβλωση της αγοράς που σέβονται τους θεσμικούς ρόλους και επιταχύνουν τις διαδικασίες και τις κάνουν πιο εύκαμπτες τις διαδικασίες. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μουσκαρντίνη και τώρα πάμε για το S&D τον κύριο Πυρίλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των, των διαφόρων ε, καταγγελιών για την ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήθηκε. Αυτό οφείλεται στην αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες χώρες ε, που αντιμετωπίζουν ε, με αυτόν τον τρόπο τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Περνάμε οικονομική και χρηματοστητική κρίση όμως 332 μέτρα προστατευτικά υιοθετήθηκαν από τους διεθνείς εταίρους ε, την τελευταία διετία. Πιστεύουμε εμείς σε διεθνές εμπόριο που είναι ελεύθερο, ισότιμο που βασίζεται σε κοινούς κανόνες που ισχύουν για όλους. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων για την υπεράσπιση του εμπορίου ε, που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη για να διορθώνουν τις καταστάσεις που δημιουργούνται από την παρανομία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τις συνέπειες που έχουν που μπορεί να έχει η μεταρρύθμιση της επιτροπολογίας όσον αυτό το εργαλείο. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές διαπραγματεύσεις, διπλωματικές διαπραγματεύσεις για να αποφασιστεί πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα anti-dumping. Αν γίνει αυτό θα αποδυναμωθεί μια διαδικασία που αντιθέτως θα έπρεπε να παραμείνει ε, ε, εδρεωμένο πάνω σε αντικειμενικά στοιχεία και κριτήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμίστες ο κύριος Σαλ Σαχραούι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που μας είπε ο κύριος Στέρντι προηγουμένως. Ε, είναι καλό υπηρέτη, αλλά όχι και Αφέντη ε, το anti-dumping. Χρησιμεύει την προστασία τη της οικονομίας, των εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ε, μπορεί ε, να γίνει κατάχρηση για λόγους προστατευτισμού με στόχο να κλείσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές, τις εξαγωγές τρίτων χωρών. Επίτροπε, σα απευθύνω έκκληση να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσετε τη χρήση μέτρων anti-dumping για προστατευτικούς σκοπούς και για το κλείσιμο των ευρωπαϊκών αγορών ε, στι στις όλου του υπόλοιπου κόσμου. Η κλειστή Ευρώπη δεν θα είναι καλή για κανέναν. Στο παρελθόν, όταν ήταν ανοιχτή και συνεργάσιμη η Ευρώπη, τελικά υποφελήθηκαν όλοι. Να το έχετε κατά νου σας, παρακαλούμε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Σαχραντήλ. Τώρα α, ο κύριος Μπιζότο δεν είναι εδώ. Οπότε περνάμε στη διαδικασία κάτσε διάει. η κυρία Κιώστιγκερ Μερσή κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι για τι αναπτυσσόμενες και αναδυόμενε χώρε το πρόβλημα του αντιντάμπινγκ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνονται συμφωνίε με τρίτε χώρε, θα πρέπει να επιμένουμε σε ρήτρε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Όταν οι χώρε δεν έχουν υψηλή ποιότητα, φυσικά βασίζονται στην τιμή για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Επομένως, εγώ βλέπω με μεγάλη ανησυχία αυτό το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο στον ΠΟΕ. Εμείς στην Τόχα δεν θα πρέπει να κάνουμε συμφωνίες οι οποίες θα επιτρέπουν το ντάμπινγκ, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πρότυπα του περιβάλλοντος και της εργασίας. Πολλέ φορέ για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση η οποία προκύπτει από το dumping, οδηγούνται στην εξαφάνιση πάρα πολλέ επιχειρήσει. Όταν κάνουμε λοιπόν και την ε, εξέταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμερική, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να τονίσει τα πρότυπα αηφορία περιβάλλοντο και κοινωνικού επίπεδου. Και χαίρομαι για αυτή την δήλωση τη Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούστιγκερ. Και τώρα για να κλείσει ο Επίτροπος Τεχούχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομη απάντηση. Έπρεπε να απαντήσω ακόμα στο ερώτημα του κυρίου Σόλτς. Όσον αφορά την περίπτωση των, των, των, του Fiberglass, σαν τον Μπαν, τους υπολογίζει ε, τι συνέπειε που θα έχει αυτό όσον αφορά τι δοκιμέ για το δημόσιο συμφέρον. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει μπορούν να συμμετάσχουν στι διαδικασίε. Ε, έχουμε μια γραμμή helpline για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να τι βοηθήσουμε στην εργασία. Όμω οι συνέπεια σε αυτή την περίπτωση ήταν μικρέ, διότι η Κίνα έχει μόνο 14% ε, τη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και το ερώτημα που έθεσε ο κ. Ζαραντίλ όσον αφορά την χρήση των μέσων πράσπιση του εμποδίου σαν προστατευτικό εργαλείο. Υπάρχει κίνδυνο να συμβεί αυτό αλλά ο κ. Ζαγραντήλ βλέπω ότι είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Ο μόνος παράγοντας επηρεάζει τον αριθμό των υποθέσεων είναι ο αριθμός των καταγγελιών που παραλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, η ποιότητα των στοιχείων που παρέχονται. Η, Ευρωπα... πολιτική πάσπιση στο εμπορίο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής... ακολουθεί κανόνες που ταιριάζουν στους κανόνε του ΠΟΕ. Αν συγκρίνεται του φακέλου και υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει dumping, ξεκινά έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το μεταξύ εξαφανίστηκε και ο κ. Ζαραντήλ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ετερματίστη η ανταλλαγή απόψεων. Η επόμενη ολομέλεια λαμβάνει χώρα στις 25 Νοεμβρίου από τις 9 ως τις 1 και από τις 3 ως τις 7. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και είναι στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό ύπνο σε όλους διότι τελείωσε η συνεδρίαση.